να κάνει μια σύντομη παρατήρηση λίγο πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο. First in this point of order. Πρόεδρε, στο ε, ως διαδικαστικό να μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά να σας συγχαρώ για την εξαιρετική ε, νίκη σας ε, ε, τον προηγούμενο μήνα ε, μετά από μια εκλογική εκστρατεία η οποία κέρδισε το σεβασμό μου προς το πρόσωπό σας και γι' αυτό ζητώ αυτό το διαδικαστικό για το σεβασμό τον οποίο σας ε, τρέφω. Ζήτησα την ε, ψήφο των συναδέλφων ως υποψήφιος πρόεδρος προκειμένου να διαφυλάξω την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού και να εξασφαλίσω ότι θα είναι πάντοτε αμερόληπτος ο πρόεδρος όπου αναφέρεται στο άρθρο αυτό ότι ο πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει το λόγο μόνο για να συνοψίσει ή να ζητεί από τους συναδέλφους να τηρήσουν την τάξη. Εάν πρόκειται να λάβει το λόγο θα πρέπει να φύγει από το Προεδρείο και να μην, το, ε, να μην ξανακαθίσει σε αυτό πριν να έχει ολοκληρώσει την ομιλία του. Ε, ύστερα από τη χθεσινή λοιπόν ε, περίπτωση με τον κύριο Φαράτζο για την παρέμβασή του, με λόγια τα οποία εγώ δεν συμφωνώ πάντα, θα ήθελα να μας διαβεβαιώσετε ότι θα τηρηθεί το άρθρο 23 έναντι κάθε ενός βουλευτού ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας και εθνικότητας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις προφορίες. Έχουμε την πρώτη έκθεση του κυρίου Σάριου Βόλσκι με μία μόνο ψηφοφορία. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την έκθεση Watson. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έκθεση ρέγνερ με ειδική πλειοψηφία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Ehrenhauser υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Σπερώνη. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να ζητήσω ηλεκτρονική επαλήθευση για την ψηφοφορία επί της έκθεσης Ρέγνερ. Δεδομένου ότι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Κύριε Σπερώνη, καταρχάς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεύτερον, σας διαβεβαιώνω ότι είχαμε ξεπεράσει κατά πολύ την ειδική πλειοψηφία. Είμαι σε θέση να το διαβλέπω αυτό ξεκάθαρα εδώ. Στην επόμενη έκθεση υπέρ Έρενχάουσεν λοιπόν κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έκθεση λένε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κατάλογο ισχυρισμό ε, διατροφής η κυρία Ζόμερ ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να κάνω μια σύντομη δήλωση, γιατί έχει επικρατήσει σύγχυση ως προς την ψηφοφορία αυτή. Εάν θέλουμε να κατα... Εάν θέλουμε να καταδικάσουμε, να απορρίψουμε δηλαδή την παραπληροφόρηση του ε, καταναλωτή θα πρέπει να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα. Εάν θέλουμε να παραπλανάται ο καταναλωτής πρέπει να καταψηφίσουμε το ψήφισμα και αυτό το λέω για να είναι ξεκάθαρο διότι πολλά ήταν τα λόμπι τα οποία προσπάθησαν να επηρεάσουν. Όποιος είναι κατά λοιπόν της παραπληροφόρησης υπερψηφίζει. Καλώς ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται υπέρ, λέει η κυρία Ζόμερ. Ich schließe die Abstimmung. Πέρας Εγκρίνεται. 393 ψήφοι καλύπτεται η ειδική πλειοψηφία που απαιτείται. Και τώρα ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ. Το παρακαλώ. Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική ψηφοφορία, φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει. Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30 Ιανουαρίου. Το συνολικό κείμενο του ψηφίσματος της ομάδας Γκούε καταρχάς. Ολόκληρο το κείμενο ΓΚΟΕ υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα το κείμενο ολόκληρο του κοινού ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατών Άλντε Πρασίνων. Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Με ονομαστική ψηφοφορία σας παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 443 ψήφοι υπέρ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την πρόταση ψηφίσματος για το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τώρα, ε, το, το κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων δυνάμει της ε, παραγράφου 3 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές επαληθεύμα Πέρας τη ψηφοφορία. Απερίφθη. Ζητώ συγγνώμη, προκαταβολικά φαίνονταν διαφορετικά από το Προεδρείο η κατάσταση. Τροπολογία υπαριθμών 2 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία. τροπολογία 3, με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται η τροπολογία παριθμών 3. Η υπαριθμών 4 τροπολογία τώρα παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Γρήγορα παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου υπαριθμών 6, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου με πρόταση για προφορική τροπολογία που θέλει να παρουσιάσει ο κύριος Πρέντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεύτερο τμήμα του εδαφίου 6. Θέλουμε να αντικατασταθεί το only από mainly. Το είπα και χτες. Χρειαζόμαστε μια πιο έντονη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Ιράν. Το ΕΛΚΑ δεν θέλει κυρώσεις ε, έτσι απλώς. Η απόφαση για κυρώσεις δεν είναι εύκολη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ιράν έχουμε πολλούς λόγους να ανησυχούμε. Πρέπει να είμαστε λοιπόν απόλυτοι και να μην αποδυναμώσουμε το μήνυμα. Απορρίπτει κανείς την υποβολή προφορικής τροπολογίας. Όχι, καλώ τότε ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. αρχίζουμε υπέρ. Με έλεγχο παρακαλώ στα κουμπιά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Υπαριθμών πέντε τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ας προχωρήσουμε. Ονομαστική ψηφοφορία για την υπαριθμό 6. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Κάρας έχει κάποια δυσκολία στην ψηφοφορία. Παρακαλώ οι τεχνικοί μας να τον ε, βοηθήσουν. Πέρα της ψηφοφορίας, απερίφθη. Τελική ψηφοφορία για το συνολικό κείμενο, στο, όπως τροποποιήθηκε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και οι λοιπές προτάσεις ψηφισμάτων των άλλων ομάδων. Ως εκ τούτου καταπίπτουν. Και τώρα κυρίες και κύριοι... Θα περάσουμε στην ψηφορία του κυρίου Φίσα Σαξιέλα, ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διάστασης του Αθλητισμού. Είναι το όνομα της εκθέσεως, τίτλος εκθέσεως. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ονομαστική ψηφορία για σχεδόν το σύνολο των τροπολογιών. Σχεδόν όλες τις τροπολογίες. Διάσταση λοιπόν του αθλητισμού. Τροπολογία μάλλον στο, στην πρώτη παράγραφο χωρί τροπολογία, αρχικό κείμενο δηλαδή, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7. Παράγραφος 7. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Εγνεκρίθη. Παράγραφος 22 ή σημείο 22. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πρέπει να σας ρωτήσω εάν μου επιτρέπετε να ψηφίσουμε ομού τις λοιπές τροπολογίες, on block. Καλώς 29 με 100. εκατό χωριστά και έτσι προτείνω το εξής να τις ψηφίσουμε χωριστά με ξεχωριστή ε, ονομαστική ψηφοφορία και τις υπόλοιπες on block παρακαλώ ομού. Λοιπόν, 29 πρώτα, η 29 άρχεται ψηφοφορία. Παράγραφος 29. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 76. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πολύ καλά. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την 100, υπαριθμόν 100 παράγραφο, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα παρακαλώ να ψηφίσουμε όλα τα άλλα, όλες τις άλλες παραγράφους μαζί. Δεν χρειάζεται να τις εκφωνήσω μία-μία.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 Ω προ τη διαδικασία και τη σειρά τη ψηφοφορία αποφασίζει ο πρόεδρο. Ε, αποφάσισα λοιπόν ότι ψηφίζουμε ομού τι λοιπέ τροπολογίε. Παρακαλώ να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Τις λοιπές παραγράφους άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται το συνολικό κείμενο τώρα υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, σας ευχαριστώ. Έκθεση Ιτήργουάης Αγγούλο. Έχουμε τις τροπολογίες 2 έως 4 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Παράγραφος 4 του αρχικού κειμένου. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχετε διαδικαστικό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε σε αυτό το σώμα, όταν ζητούνται ονομαστικές πληροφορίε από όλες τις πλευρές, από όλες τις ομάδες και όλα τα κόμματα, τείνουμε να σεβόμαστε τα αιτήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι είστε νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, το να αποφασίζετε αυθαίρετα για απλό ψηφοφορία είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ε, μπορεί, Πρόεδρε, να κάθεστε εκεί με ψήφους, ε, λίστες ψηφοφορίας των σοσιαλιστών ή του ΕΛΚ. Υπάρχουν άλλες ομάδες όμως σε αυτό το σώμα που θέλουν να ψηφίσουν με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι εάν εγώ έχω ένα κατάλογο ψηφοφορία από την ομάδα μου και έχουμε ζητήσει μέσω τη φυσιολογικής διαδικασία σωστά και εγκαίρω ονομαστική ψηφοφορία που τυχαίνει να είναι κατά τμήματα και αν δεν συμφωνούμε να τις ε, ψηφίσουμε unblock, όπως μπορεί να μην συμφωνούν ούτε και άλλοι συνάδελφοι από άλλες ομάδες, ε, θα πρέπει αυτό να γίνεται. Πιστεύω πως κάνατε λάθος και ελπίζω πως στο μέλλον θα συνεχίσετε με σωστό και δημοκρατικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Μη μου φωνάζετε, Πρόεδρε, μη μου φωνάζετε. Σας κατενόησα. Σας κατανόησα διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία και η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ζήτησε ψηφοφορία ομού. Πράγμα και το οποίο δέχθηκα. Τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία μας στην έκθεση του Ργάης Άγγουλο. Παρακαλώ, πέντε. Κατά αποχές. Στο δεύτερο τμήμα της ονομαστικής ψηφοφορίας άρχεται. Με ονομαστική ψηφοφορία, μάλλον άρχεται. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπο... 33, ε, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα και πάλι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. στο ε, αιτιολογικό ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφορία. πέρας, εγκρίνεται. F, σίγμα ταφ, άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται θεολογική σκέψη AQ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Σε δύο τμήματα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της ίδιας παραγράφου. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της AQ. Πέρασε Εγκρίνεται. AT, ε αιτιολογική σκέψη AT, ε υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. AX, ε πρώτο τμήμα, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το όλο κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κύριε Άτκινς. Πρόεδρε. Θέλω τη συμβουλή σας για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Πρώτον, συγχαρητήρια που ξεκινήσατε στην ώρα σας και προσπαθείτε να προχωρήσουμε γρήγορα με ευγνώμων σε εσά που ακούτε. Αλλά πώς εξηγείτε είτε στη δίκηση, είτε πώς να εξηγήσω εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια ότι εγώ ζητάω μια σειρά ονομαστικών ψηφοφοριών και θέλω να ψηφίσω υπέρ σε ορισμένε και κατά στι άλλε. Και εσεί βάζετε σε ψηφοφορία όλε μαζί. Οπότε πώ θα μπορέσω εγώ να υπερψηφίσω, να καταψηφίσω διαφορετικά. Εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια αυτό πώ θα το εξηγήσω. Και πώ θα το εξηγήσω και στην δίκηση όταν του πω ότι εγώ ήθελα σε άλλε να ψηφίσω υπέρ, σε άλλε κατά και σε άλλε να κρατήσω θέση αποχή. Okay. Ο Πρόεδρος, κύριε Άτκινς, όταν έχουν ε, ετίματα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία, πρέπει να τα θέσει δυνάμει της 166 παραγράφου 5 διατάξεως του κανονισμού σε ε, ψηφοφορία χωριστά δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά μπορεί να ζητήσει από, την, ε, από το σώμα την γνώμη του, την άποψή του για το αν μπορεί on ο ομού δηλαδή, να ψηφίσει τις τροπολογίες. Σας διαβάζω λοιπόν το κείμενο. Παρακαλώ, ακούστε με, πρόκειται για το κείμενο του κανονισμού. Ο Πρόεδρος μπορεί άλλες και συμπληρωματικές τροπολογίες να τις υποβάλει ομού σε ψηφοφορία. Πρόκειται για τη διαδικασία της παραγράφου 5, όπου ερωτώ την Ολομέλεια το σώμα εάν συμφωνεί πράγμα και το οποίο έπραξα και αν εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε τέτοιες τροπολογίες να τις έχω θέσει ψηφοφορία χωριστά μία-μία, τότε να με ενημερώνετε στην διάσκεψη των Προέδρων, έτσι ώστε την κάθε μία τροπολογία να την ψηφίσουμε χωριστά. Θεώρησα ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο να κάνουμε τη δουλειά μας πιο αποτελεσματικά. Εάν όχι, να το συζητήσουμε. Περνώ τώρα στην έκθεση Μπάστος, προ, ε, πρόγραμμα Δάφνη, παράγραφος 8 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 15, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη ΚΑΠΑ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου, παρακαλώ. Κάποιος να με βοηθήσει. Καλώ, θα σα ε, στείλουμε ένα τεχνικό για υποστήριξη. Και τώρα στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση Μπάστο με ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ, άρχεται. Ja. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Μπάστος. Um, Ευχαριστώ. Στην επόμενη ψηφοφορία υπάρχουν λίγες εδώ και αντί να σηκώνουμε το χέρι συνέχεια, μήπως θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, παρακαλώ, αν μπλοκ. Έκθεση Νικολάη. Παράγραφος 4, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4, πρώτο, η Παύλα, υπέρ. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της πρώτης Παύλας, υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Σημείο 4. Δεύτερη παύλα. Πρώτο τμήμα. Περ, κατά. Αποχές. Στα ελληνικά ο πρόεδρος. Εγκρίνεται στα ελληνικά ο πρόεδρος. Παραγράφος 4-3. Τρίτη παύλα δηλαδή. Συγγνώμη, 4-2 διορκώνει ο πρόεδρος, δεύτερη παύλα, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. τρίτη παύλα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τρίτης παύλας υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεκαεπτά. τέταρτη παύλα, υπέρ, πρώτο τμήμα, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 30 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και τώρα το σύνολο του, του κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε τη έκθεση του κυρίου Νόιζερ Παράγραφος παριθμών 11, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα του 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 Μάλιστα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 21 στο δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το 26, δεύτερο τμήμα. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια. Έκθεση Σμιτ. Ετήσια έκθεση για τη φορολογία, δεύτερη παράγραφος, πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόλυτη αναρχία επικρατεί στην ψηφοφορία υπέρ του πρώτου τμήματος κατά τώρα αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την παράγραφο 8 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο υπαριθμών 8. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παραγράφος 9 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγράφος 11 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 50. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το όλο κείμενο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση ΣΦΑΠ, ετήσια έκθεση για την ε, πολιτική ανταγωνισμού έχουμε μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων, ΙΣΙΑΡ Πρασίνων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ και έτσι τέλειωσε η ψηφοφορία. Vielen Dank. Waren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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Έχω να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μου γνωστοποίησαν την κατάσταση, την αντικατάσταση του κυρίου Μιχαήλ Τρεμόπουλου από τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο με ισχύ από την Δευτέρα Φεβρουαρίου 2012. Καλωσορίζω λοιπόν τον νέο συνάδελφο και υπενθυμίζω ότι δυνάμη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως ότου ελεγχθεί η εντολή ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο και του ευχόμαστε καλή θητεία. Επίσης, έχω λάβει από τις ε, ομάδες PPE, S&D, VER, ALDE, ECR, GUE και EFD τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Στην Επιτροπή Ίντα, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η κυρία Μαρία Μπαντία Ικουτσέ στη θέση του κυρίου Εμίλιο Μενέντες Δελβάλε. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, Budget, ο κύριος Ρίτσαρτ Ashworth στη θέση του κυρίου Λάγιος Μπόκρος. Έμβη, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ο κύριος Λάγιος Μπόκρος στη θέση της κυρίας Τζούλη Γκίρλινγκ. Τραν, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ο κύριος Φίλιπ Μπράτμπουρν στη θέση του κυρίου Ρίτσαρτ Τσαρνέτκι. Ρέτζι, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Ρίτσαρτ Τσαρνέκη στη θέση του κυρίου Φίλιπ Μπράτμπουρν. Με συγχωρείτε, ε, στην Επιτροπή Ρέτζη, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, αναλαμβάνει καθήκοντα επίσης ο νέος συνάδελφος, ο κύριος Νικόλαος Χρυσόγελος. Άγκρη, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου, η κυρία Τζούλι Γκέρλιν στη θέση του κυρίου Ρίτσαρτ Άσουορθ. Καλτ, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Ο κύριος Εμίλιο Μενέντες Δελβάλε στη θέση της κυρίας Μαρία Μπαντία Εκουτσέ. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ορβηγία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ο κύριος David Campbell Bannerman στη θέση του κυρίου Σαΐτ Καμάλ. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο ο κύριος Σαλβατόρε Ταταρέλα στη θέση του κυρίου Ποτίτο Σαλάτο. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν ο κύριος Ποτίτο Σαλάτο στη θέση του κυρίου Σαλβατόρε Ταταρέλα. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Η κυρία Ινιές Κριστίνα Τζουμπέρ. Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Ο κύριος Ταντέους Σιμάνσκι δεν είναι πλέον τακτικό μέλος. Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ευρωπαϊκής ένωσης αρμενίας ευρωπαϊκής ένωσης αζερβαϊτζάν και ευρωπαϊκής ένωσης γεωργίας ο κύριος Γεώργιος Παπαστάμκος στη θέση του κυρίου Ιωάννη Τσουκαλά αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλά στη θέση του κυρίου Γεωργίου Παπαστάμκου αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης άκε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γιάτζεκ Όλτζερ Κούρσκι στη θέση του κυρίου Ορέστε Ρώση. Και τέλος, αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρώπης Λατινικής Αμερικής, ο κύριος Ταντέους Τσιμάνσκι δεν είναι πλέον τακτικό μέλος. Επίσης, έχω λάβει από το Συμβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το σκεπτικό που το οδήγησε στην έγκρισή της, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης. Η προθεσμία των τριών μηνών, την οποία διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφανθεί, αρχίζει συνεπώς από αύριο, 3 Φεβρουαρίου του 2012. θέση του Συμβουλίου εν ώψη της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών υπαριθμών 1290 του 2005 και υπαριθμών 1234 του 2007 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Και πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φόξ Άσλεϊ. Ο κύριος Φόξ Άσλεϊ είναι στην αίθουσα. Προχωρώ στον επόμενο γορητή, η κυρία